και έχω μία ανακοίνωση για την επόμενη συζήτηση. Ο Πρόεδρος έχει βάλει έτοιμα τροποποίησης της Επιτροπής ε, από το ΕΛΚ και το ΙΕΝΕΦ. Αυτό θα παρουσιαστούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στην υιοθέτηση του